Η ημερήσια διάταξη προβλέπει δηλώσει του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επισκόπηση τη Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Να θυμίσω σε όλου του συναδελφού ότι για τη συζήτηση αυτή προβλέπεται διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Δεν προβλέπεται μόνο διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και δεν θα γίνουν δεκτέ και ε, δεκτά αιτήματα γαλάζια κάρτα. Πριν δώσω το λόγο στον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κούρτ, να ευχαριστήσω την Αυστριακή Προεδρία για την εντατική συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Θα ευχαριστήσω επίσης την Αυστριακή Προεδρία για την πρόσκληση προς το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετάσχει στην ε, εκδήλωση για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, τη Σχετική Σύνοδο, όπου συμμετείχαν και ο πρόεδρο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τούσκ, και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η όλη σύνοδο. Ευχαριστώ του εκπροσώπου και τη Αυστριακή κυβέρνηση που συμμετείχαν στι ε, συνόδου του Κοινοβουλίου και σα ευχαριστούμε και για την έλευσή σα στι Βρυξέλλε. Με όλε αυτέ τι ευχαριστίε, δίνω το λόγο στον Κακελάριο Κούρτ. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, κύριες και κύριοι πρόεδροι των ομάδων και βουλευτές. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της Αυστριακής Προεδρίας. Έχουμε πίσω μας έξι εντατικούς μήνες, ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα εργασίας και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα αυτής εξ αρχής να αναφέρω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Κομισιών. Και σας ευχαριστώ για την στήριξη στην Προεδρία μας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας πάντα αποδίδω μεγάλη σημασία στην συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Μπόγνα Στράους ε, και την Καρολίνα Ερστάτλερ, τις υπουργού που μας εκπροσώπησαν στις ημέρες της Ολομέλειας. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω και για τους 161, ε, τις 161 διμερείς συναντήσεις στα πλαίσια του διαλόγου που είχαμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν Συμβούλιο Κοινοβουλίου και Κομισιόν για την διάθεση συμβιβασμού που επέδειξαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της Αυστριακής Προεδρίας, ε, τον πρέσβηρά μας, ε, τον Αλεξάνδρ Σάινμπεργκ και τους άλλους της ε, Βρυξέλλες και βεβαίως ε, επειδή κάθε προεδρία είναι μόνο ένας κρίκος στην αλυσίδα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους στο τρίο την Εστονία και την Βουλγαρία και με της ευκαιρίας ε, για να ευχηθώ κάθε επιτυχία και στην Ρουμανική Προεδρία. Κυρίες και κύριοι, είχα έρθει εδώ και τον Ιούλιο και τότε είχα πει πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το αυτονόητο και θα πρέπει καθημερινά να προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Και επειδή είχαμε και δύσκολες συζητήσεις, είχα πει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα που μας ενώνουν από όσα μας χωρίζουν. Και τα ίδια θα έλεγα και σήμερα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την πρόκληση της πολύ πολύπλοκης δομής λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν όμως παρόλα αυτά πολλά πράγματα που μας ενώνουν ε, και μπορούμε να συνεργαστούμε για να τα λύσουμε. Ώστε δεν υπάρχει καμία εναλλακτική σε αυτήν την συνεργασία και στην διάθεση να βρούμε συμβασμούς. Χαίρομαι για το ότι τους προηγούμενους έξι μήνες ε, καταλήξαμε σε κάποιους συμβιβασμούς και έτσι ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να έκανε κάποια βήματα στην σωστή κατεύθυνση σε πολλά ζητήματα. Δεδομένης της συγκυρίας, θα ήθελα να αναφερθώ στο Brexit και τις σχετικές προκλήσεις. Όταν αναλάβαμε την Προεδρία τον Ιούλιο, είχαμε την απέτηση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την Ευρώπη των 27. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Κομισιόν και τον Μισελ Μπαργιέ για τις διαπραγματεύσεις, γιατί καταφέραμε και με την δική μας στήριξη να διατηρηθεί η ενότητα των 27 και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν ε, μπορεί να κατηγορηθεί για τίποτα στις διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Διαπραγματευτήκαμε μια ισορροπημένη πρόταση και διασφαλίσαμε και τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Ακόμα και αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα της απόψινής ψηφοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία και οι επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι, ελπίζω να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι οι 27 και να έχουμε μια κοινή στάση Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Η Αυστρία οπωσδήποτε θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει αυτή τη γραμμή. Εκτός από το Brexit έχουμε μια Ευρώπη ε, που εστίασε σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια και η καταπολέμηση της παράνομης ε, μετανάστευσης, ε, δεύτερον η εφημερία και τρίτον η γειτονία. Και βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την σταθερότητα στη γειτονιά μας. Για το πρώτο θέμα, την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Παρά το μπλοκάρισμα που υπήρξε στο θέμα της κατανομής, επετεύχθη κάποια πρόοδο στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ειδικά με την Αίγυπτο, αλλά και με άλλες χώρες, καταφέραμε να διασφαλίσουμε πως η διάσωση δεν θα γίνεται μόνο από ευρωπαϊκά σκάφη ε, που συνδέεται με ένα άμεσο εισιτήριο προς την Ευρώπη, αλλά να υπάρξει διάσωση και από την Αίγυπτο, την Λιβύη και άλλους. Και μετά την διάσωση οι άνθρωποι να επιστρέφουν στη Βόρεια Αφρική. Αυτό οδηγεί στο ότι συνολικά σήμερα έχουμε 95% λιγότερες αφήξεις στην Ευρώπη από το 2015 και το σημαντικό είναι όχι μόνο η μείωση των αφήξεων αλλά και των θανάτων που μειώθηκαν δραματικά σήμερα η κεντρική οδός η μεσογειακή της Ιταλίας de facto έχει κλείσει τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχαμε καθόλου αφήξεις καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία των Υπουργών εσωτερικών για την εντολή της Frontex ε, να συνεργάζεται με τρίτες χώρες αλλά να έχει και ένα σημαντικότερο ρόλο και όσον αφορά την ε, ενίσχυσή της με προσωπικό εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν και θα ήθελα να ζητήσω και από σας μιλήστε με τους αρχηγούς των κυβερνήσεών σας, με τις κυβερνήσεις σας. Υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να πιστούν. Όσον αφορά το θέμα της κατανομής. Προσπαθήσαμε να μην επιμείνουμε, αλλά να φέρουμε μία νέα πρόταση. Την υποχρεωτική, αν θέλετε, αλληλεγγύη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις θετικές της κουβέντες. Για το θέμα της ανταγωνιστικότητας, της ευημερία, την βιωσιμότητα του οικονομικού χώρου που λέγεται Ευρώπη. Ε, δώσαμε βάρος ε, στην βιωσιμότητα της εσωτερικής αγοράς και χαίρομαι για το ότι είχαμε κάποιες ε, θετικές πρόοδους στο θέμα της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς όπως παραδείγματο χάρη το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον ετέθη το ζήτημα της φορολόγησης των ε, γιγάντων του διαδικτύου. Έχει υπάρξει μια μεταβολή των απόψεων εντός του Συμβουλίου. Βεβαίως δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι αποφάσεις και θα ήθελα και πάλι να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε να πείσουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι ακόμα επιφυλακτικές. Για την αηφορία, ε, αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερο ως Αυστρία και χαίρομαι για το ότι υπήρξε απαγόρευση κάποιων χημικών ουσιών, αλλά βεβαίως συμφωνήσαμε και στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα ΙΟΤΑΧΗ, μια μεγάλη επιτυχία Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν. ένα αποτέλεσμα του Τριμερού διαλόγου. Η προστασία στο χώρο εργασίας για, από κάποιες ε, καρκινογόνες ουσίας επίσης, ε, ουσίες με συγχωρείτε, και η σχετική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είναι κάποια βήματα που θα ήθελα να αναφέρω. Μια πραγματικά ισχυρή Ευρώπη, μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται και έναν σύγχρονο προϋπολογισμό και ομολόγο. πως οι διαπραγματεύσεις ε, αυτές ε, για το ΠΔΠ ξεκίνησαν έτσι ώστε στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός ε, γι' αυτό Είχε δίκιο εδώ ο πρόεδρος της Κομισιόν ότι έπρεπε να μπούμε με ορμή στις διαπραγματεύσεις και τελικά είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι ε, περιμέναμε. Και χαίρομαι ε, για το ότι θα ολοκληρωθούν προσεχώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις ε, κατόπιν. Έχουμε την πολιτική γειτονίας Εκεί ως Αυστριακός βεβαίως ε, είμαι ευγνώμων για το ότι τελικά καταλήξαμε στο να εστιάσουμε σε μια ενίσχυση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Είχαμε μια επίλυση του θέματος ε, του ονόματος ε, και ε, ανοίξαμε κάποια κεφάλαια με την Σερβία και το Μαυροβούνιο, κάτι το οποίο δείχνει πως υπάρχουν προοπτικές για αυτήν την περιοχή. Και χαίρομαι για το ότι η Ρουμανία και προσεχώς η Βουλγαρία θα δώσουν ιδιαίτερο βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. τον πρόεδρο Ταγιάννη. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το φόρουμ για την Αφρική που είχαμε στην Βιέννη με την Αφρικανική Ένωση όπου προσπαθήσαμε να δούμε τα ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης της Αφρικής και να μην παραδώσουμε αν θέλετε την Ήπειρο αυτή στους Κινέζους κυβερνήσεις ε, είχαν πάρα πολύ καλές επαφές και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους κατέστησαν δυνατό αυτό το φόρουμ. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο αφορά και είναι σημαντικό για εμάς στην Αυστρία ε, για ιστορικούς λόγους, ε, την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού είχαμε κάνει μια διάσκεψη στη Βιέννη με όλες τις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης ε, και καταλήξαμε και σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων γιατί δεν είναι δυνατόν οι Εβραίοι στα διάφορα κρατημένα να μην αισθάνονται ασφαλείς και πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, τον Πρόεδρο Γιούνκερ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως ε, τον Πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη, αλλά και τους άλλους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων για την καλή και επικοδομητική συνεργασία. Προσπαθήσαμε πάντα να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς για να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταλήξουμε σε συμβασμούς και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χαίρομαι για το ότι καταφέραμε κάποια πράγματα σε κάποιους τομείς και δεσμεύουμε ότι ως Αυστρία θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια που υπάρχει κάποιο άρωμα προεκλογικού αγώνα σε όσους θα είναι υποψήφοι τον Μάιο να ευχηθώ καλή επιτυχία και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Ελπίζω όμως αυτή η συζήτηση να γίνει πάντα με σεβασμό στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και όπως θέλουν και οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία τους έξι αυτούς μήνες και καλή επιτυχία εύχομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, Chancellor, Σας ευχαριστούμε, Καγκελάριε, για την ομιλία σας, αλλά και για την ε, σαφή ε, δέσμευσή σας και αφοσίωση να καταπολεμήσετε τον αντισημιτισμό. Είναι ε, σημαντική προτεραιότητα η ανεξιθρησκεία και ο διαθρησκειακός διάλογος για αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας, λοιπόν. Σα ευχαριστώ. Και τώρα ο Πρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζαν Κλόντ Γιονκέρ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σα, μποντζόρνο, Κύριε και κύριοι βουλευτέ, κύριε Καγκελάριε, κυρία Υπουργέ και λοιποί. Υπουργοί, κύριε Πρέσβη, ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της Αυστριακής Προεδρίας οφείλεται σε εσά. Δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα όσα είπε ο Καγκελάριος. Ο απολογισμός της Αυστριακής Προεδρίας είναι εντυπωσιακό. Αν δει κανείς τον αριθμό των συμφωνιών στις οποίες κατέληξαν Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν 134 θέματα είχαν επιτυχή κατάληξη και τα μισά από αυτά με το Συμβούλιο και τα μισά με το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, και συγκρίνω αυτά τα οποία κατάφερε η Αυστριακή Προεδρία με αυτά τα οποία κατάφεραν άλλες προεδρίες ε, από τις οποίες είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και θεωρώ ότι ο απολογισμός είναι ε, πραγματικά εντυπωσιακό με μια σημαντική εξαίρεση. Εγώ θα ήθελα η Αυστριακή Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτήν την αδυναμία στο θέμα του Συμφώνου Μετανάστευσης του ΟΗΕ και να το συνυπογράψει. Ο Σεμπάστιαν το γνωρίζει του το έχω πει ότι θα ήταν επιθυμητό η Προεδρία του Συμβουλίου να κάνει ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση αντί να στέλνει αρνητικά μηνύματα. Αλλά γεγονός είναι επίσης ότι η Αυστρία δεν είναι η μόνη χώρα που απέρριψε αυτό το σύμφωνο. Δεν το αντιλαμβάνομαι αλλά με την εξαίρεση αυτή όπως είπα αυτή τη στιγμή αδυναμίας δεν ε, μπορώ πραγματικά να προσάψω τίποτα στην Αυστριακή Προεδρία γιατί παρά τις κάποιες ε, προκαταλήψεις ε, που υπήρχαν Ε, υπηρέτησε θα έλεγα την ευρωπαϊκή υπόθεση με μεγάλη συνέπεια, ε, συνέχεια και σοβαρότητα. Και πραγματικά απίλαυσα το πώς εμείς ως ε, Κομισιόν είχαμε πάντα απέναντί μας την ετοιμότητα της Αυστριακής ε, Προεδρίας να εγγυηθεί την ενότητα των 27 όσον αφορά τον Brexit, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ε, η συζήτηση αυτή δεν ήταν μόνο στο επίπεδο των αρχηγών κρατών, αλλά και στο επίπεδο των ειδικών. Εκεί πέρα χάραξε ξεκάθαρες γραμμές η Αυστρία και πραγματικά της αξίζει κάθε έπαινος. Είμαι ιδιαίτερος ε, ικανοποιημένο ε, για το ότι υιοθέτησε η Αυστριακή Προεδρία τις προτάσεις μας για την διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων. Εδώ πέρα πρέπει να αναγνωρίσω πως η Κομισιόν βασίστηκε στην πρόταση της αυτή στα όσα είχε προτείνει ο Αυστριακός Καγκελάριος. Γιατί είχε πει ότι μέχρι το 2000 ένα έτος θα πρέπει να έχουμε 10.000 ε, άτομα προσωπικό και διαπιστώνουμε τώρα ότι ο Αυστριακός ε, Καγκελάριος ε, και ο Πρόεδρος Κομισιόν ήταν οι μόνοι που επέμεναν σε αυτό το οποίο όλοι ήθελαν και προσπάθησε η Αυστριακή Προεδρία να προωθήσει και να διατηρήσει ζωντανή αυτή την ιδέα. Παρατηρείτε ότι με ταλαιπωρεί ο λαιμό μου, κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει ότι δεν θα με υποστείτε για πολύ. Οπότε θα ήθελα να ξεκαθαρίσω την διγλωσία του Συμβουλίου. Δηλαδή, μα ζητάνε όλοι να κάνουμε κάτι για την προστασία των συνόρων. Κάνουμε κάτι σε συνεργασία με τον Καγκελάριο και μετά έχουμε διάφορε ε, παραπλευρές ε, κινήσεις. Ε, είτε τηρούμε τα συμφωνημένα και αυτά που μας ζητάνε ή καλύτερα να μην μιλάνε κάποιοι. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον ε, και την Αυστριακή Προεδρία για τη στήριξή τους. Και ε, σας είπα ότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις ε, που υπήρχαν, προωθήθηκε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνομιλία στην καγκελαρία και σας είχα παρακινήσει να το προωθήσετε. Το έκανε η Αυστριακή Προεδρία παρά τις επιφυλάξεις που είχε και είμαι ευγνώμων ε, για το ότι επιτέλους μετά την αρχή των τραπεζών έχουμε και μια αρχή ε, για την εργασία. Γιατί είναι λάθος η αίσθηση ότι η Ευρώπη στρέφεται κατά του εργαζόμενου. Όποιος προστατεύει τις τράπεζες πρέπει να προστατεύσει και τους εργαζόμενους και εδώ πέρα μας βοήθησε πολύ η Αυστριακή Προεδρία για το πί δημοσιονομικές προοπτικές. Πραγματικά και εδώ πέρα οφείλουμε να επενέσουμε και να αναγνωρίσουμε την Αυστριακή Προεδρία. Κατάφερε λοιπόν κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια να πραγματικά φτιάξει έτσι τα διαπραγματευτικά κουτιά όπως ε, λέγονται έτσι ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να έχουν μια διαπραγματευτική βάση που τους επέτρεψε στα θέματα των δημοσιονομικών προοπτικών να επιτύχουν την πρόοδο που χρειάζεται έτσι ώστε τον Οκτώβριο και εδώ πέρα πραγματικά τα κατάφερε η Αυστριακή Προεδρία εγκαίρως να ε, καταλήξουμε κάπου. Οπότε μόνο επένους και εδώ για την Αυστριακή Προεδρία γνωρίζετε πόσο δύσκολα είναι αυτά τα θέματα με τα κουτιά αυτά και τη συναρμολόγησή τους κατάφερε λοιπόν η Αυστριακή Προεδρία να κάνει έτσι τα πράγματα ώστε να προωθηθούν και να σημειωθεί κάποια πρόοδο στις μουσιονομικές προοπτικές. Σας ευχαριστώ και για αυτά τα οποία είπατε για τον αντισημιτισμό δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα φοβόντουσαν οι Εβραίοι συμπολίτε μα να εκδηλώσουν την πίστη τους και η Αυστρία έχει κάποιους ιδιαίτερους λόγους να λέει λόγια σταράτα στο θέμα αυτό ήμουνα και στην Βιέννη από κάποιους μήνες επισκέφθηκα και την εβραϊκή κοινότητα της Βιέννης για να δείξω ότι δεν υπάρχει χώρος ε, για αντισημιτισμό και ρατσισμό στην Ευρώπη. Και στην πράξη νομίζω ε, έδειξε η Αυστριακή Προεδρία ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να καταπολεμηθεί, καταπολεμηθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Επίσης, είμαι ευγνώμων για την πρωτοβουλία για την Αφρική. Έτσι όπως λέμε σε ωραία γερμανικά υπήρξε μια, ένα high level group, μια συνάντηση υψηλού επίπεδου στην Βιέννη με τους Αφρικανούς ομολόγους μας ε, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια διασφάλιση του αφρικανικού μέλλοντος. Αλλιώς δεν θα υπάρξει διασφάλιση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Αυτό ήταν λοιπόν το σημαντικό μήνυμα της Αυστριακής Προεδρίας ε, προς την Αφρική. Και ήταν πολύ σημαντικό. Συνολικά λοιπόν, με την εξαίρεση που ανέφερα, είχαμε μια επιτυχημένη Προεδρία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο, την κυβέρνηση, τον πρέσβη για τα όσα έκαναν και τις επιτυχίες που στην αρχή της Προεδρίας δεν νομίζαμε ότι θα συμβούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν να περάσουμε στου εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ε, παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευση, γιατί όπω ε, ξέρετε έχουμε και την παρενική συνεδρίαση για την 20η επέτειο του ευρώ. Τώρα ο κύριο Βέμπερ, που είναι πρόεδρο ε, του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Καγκελάριε, κύριε Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στον απολογισμό τη προεδρία του Συμβουλίου και εμείς ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για, την για τον εντυπωσιακό αυτό απολογισμό της ε, Προεδρίας σας για τα όσα καταφέρατε αυτούς τους έξι μήνες για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ειλικρινά σας λέω, καμιά φορά είναι κρίμα το ότι οι δημόσιες συζητήσεις για την Ευρώπη αφορούν πάντα τις κρίσεις, πάντα τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν καταφέρνουμε να συζητήσουμε τα θετικά τα όσα καταφέρνουμε, αυτά τα οποία ενισχύουν την Ευρώπη. Είναι κρίμα. Έτσι, ε, βεβαίως ε, ζούμε ως πολιτική, αλλά αυτό το αποδεικνύει ιδιαίτερο η Αυστριακή Προεδρία. Ο πολιτικός απολογισμός ήδη έγινε. Ως ομάδα του ΕΛΚ θα θέλαμε να τονίσουμε τα θέματα της ασφάλειας, το Ταμείο Άμυνας, ε, ο τομέας των μη επανδρομένων αεροσκαφών επίσης ε, προσφέρει ε, πάρα πολλές ε, προοπτικές. Έχουμε το θέμα της ευημερία. Επιτύχαμε εκεί πέρα σημαντικές προόδους. Τον έλεγχο των επενδύσεων κατ' σημαντικό. Η συμφωνία με την Ιαπωνία επίσης έκλεισε και όσον αφορά τις χρεώσεις περιαγωγής, ε, το καταφέραμε όπως επίσης και για τα τραπεζικά εμβάσματα και την απαγόρευση των πλαστικών και το διοξίδιο του άνθρακα. Είχαμε αρκετές επιτυχίες ε, και αν μπορούσαμε να το μεταδώσουμε αυτό στον κόσμο θα πήγαινε και καλύτερα η Ευρώπη. Σημαντικό είναι επίσης το ότι ξεκίνησαν πολιτικές ε, συζητήσεις γιατί βεβαίως είναι κάποια διαχείριση η Προεδρία αλλά πρέπει να δώσει και κατευθύνσεις στο πρώτο άτυπο συμβούλιο στο Σάλτσμπουργκ ετέθη το ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Για εμάς είναι κεντρικό ζήτημα, είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στον τομέα της μετανάστευσης. Το θέμα της δικαιοσύνης με τον ψηφιακό φόρο. για να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί και οι μεγάλη όμιλη του διαδικτύου. Σας συγχαίρω λοιπόν γι' αυτό. Αυτό νομίζω ωφέλησε την Ευρώπη και η συζήτηση βεβαίως θα ανέφερε ο Ζανκλοντ Γιούνκερ για το εάν είμαστε στην Ευρώπη σε μια ήπειρο που μιλάμε ξανά σοβαρά για βία κατά των Εβραίων πρέπει αυτό να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα το θέμα δηλαδή του αντισημιτισμού και αυτά τα οποία μας είπαν οι εβραϊκές ενώσεις πρέπει να μας ανησυχήσουν. Και το βασικό μήνυμα εδώ πέρα είναι ποτέ ξανά. Σας συγχαίρω λοιπόν. Τέλος θα ήθελα να πω πως η Αυστρία είναι οπωσδήποτε ισχυρή χώρα με μια ισχυρή κυβέρνηση και οι πολίτες ε, νομίζω το είδαν όπως και εγώ ότι ήταν υπερήφανοι που είχαν για ένα εξάμεινο την Προεδρία της Ευρώπης ε, και ήταν ε, πάρα πολύ θετικό και αυτό το οποίο παραμένει είναι η επικοδομητική συνεργασία, η ηγεσία που επιδείξατε και η συνένεση που οδηγούν όλα αυτά σε πρόοδο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ροντρίγκε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρη, η Αυστριακή Προεδρία ξεκίνησε με ένα σημαντικό μότο, μια Ευρώπη που προστατεύει. Και πράγματι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να προστατεύει. Όμως θεωρούμε την, ότι η Αυστριακή Προεδρία παρουσίασε περισσότερα αποτελέσματα, μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη φόβων ε, και μια Ευρώπη επαναχωρήσεις και εγωισμών ε, και το λυπούμαστε γι' αυτό γιατί χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με μεγάλες φιλοδοξίες έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε και την απαραίτητη αλληλεγγύη. Αυτό ξεκίνησε με τη δραματική κατάσταση για τους πρόσφυγες. Θα μπορούσαμε να είχαμε ταχείες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής ασύλου. Όμως ε, είδαμε διάφορα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο και λυπούμαστε γι' αυτό. Η Ευρώπη θα πρέπει να καθορίσει μια πλήρη πολιτική για το μεταναστευτικό για να μπορεί να διαχειριστεί τη μετανάστευση, μια έφτακτη μετανάστευση, γιατί χρειαζόμαστε τη μετανάστευση. Αντιθέτως όμως μπλοκάρουμε κάποια κύρια τμήματα αυτής της μεταναστευτικής πολιτικής και κατόπιν. Λυπούμαστε για το τι συνέβη με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, γιατί επικυρώθηκε από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και είδαμε ότι στο Μαρακές κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κυρώνουν το σύμφωνο αυτό από την ηγεσία της αυστριακής κυβέρνησης. Και πάλι εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτό και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Όμως αυτή η έλλειψη φιλοδοξίας και αλληλεγγύης έχει συνδεθεί και με τους πολίτες. Γιατί για να δούμε τι γίνεται με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία που έχουμε. Η Αυστριακή Προεδρία θα μπορούσε να έχει παρουσιάσει ταχύτερα αποτελέσματα για όλο το σύνολο των οδηγιών που είναι απαραίτητε για την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν δυνατό η Αυστριακή Προεδρία να αναβάλει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών. Βιαζόμαστε, κύριε Καγκελαρή, για να εφαρμόσουμε αυτόν τον πυλώνα και να τον καταστήσουμε πραγματικότητα. Και κατόπιν έχουμε τις σημαντικές διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ναι, είναι κάτι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις στην Ευρώπη, και για να έχουμε και ισχυρή δέσμευση Ω προ τη συνοχή, απογοητευτήκαμε που το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι η τελική συμφωνία θα πρέπει να ληφθεί, να γίνει τον φθινό, το φθινόπωρο. Έχουμε τις προϋποθέσεις να καταλήξουμε σε μια βασική συμφωνία νωρίτερα. Και δεν κατανοούμε γιατί η Αυστριακή Προεδρία δεν ήταν ικανή να παρουσιάσει ένα πιο φιλόδεξο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Κατόπιν, είχαμε μια άλλη ευκαιρία για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Πρόκειται για κάτι που περιμένουμε εδώ και χρόνια. Η λύση είναι επιτάπητος. Μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία που θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και να δημιουργήσουμε ένα προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Κάτι που έχουν όλε οι νομισματικέ ενώσει ε, παγκοσμίω. Έχουν προπολογισμό. Όμω και πάλι η Αυστρική Προεδρία δίσταζε. Και αυτό είναι ένα ε, ζωτικό στοιχείο για να έχουμε εκ νέου συνοχή στην Ευρωζώνη και να καταπολεμήσουμε τις αποκλίσεις ε, σε αυτό το σημαντικό τομέα του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και κατόπιν φορολογική δικαιοσύνη. Ναι, χρειαζόμαστε ένα νέο ψηφιακό φόρο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα πρέπει ταχύτερα να τον υλοποιήσουμε. Έτσι, λοιπόν, από τη δική μας σκοπιά, κύριε Καγκελάρε, η Αυστριακή Προεδρία έχασε κάποιες ε, σημαντικές ευκαιρίες για να οικοδομήσει μια πιο ισχυρή Ευρώπη που χρειαζόμαστε αυτή τη συγκεκριμένη, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία. Γιατί βλέπουμε μια νέα κίνηση ιδεών και ε, βλέπουμε εδώ ότι ε, βλέπουμε εγωισμούς, ε, ακροδεξιά κινήματα και εγκλωβισμούς και απέναντι σε αυτό έχουμε την εξή επιλογή, είτε θα συμμαχίσουμε μαζί τους και θα κάνουμε κάποιες εκχωρήσεις στα κίνηματα αυτά ή θα παρουσιάσουμε μια πλήρη εναλλακτική, μια ισχυρή φιλόδοξη Ευρώπη που να μπορεί να παρέχει αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς, θεωρούμε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες και θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα νέο στάδιο που ε, τέτοιε ηγεσίε θα αναδυθούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το δικό μα μότο, κύριε Πρόεδρε. Επόμενο για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο Ζάχραντιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπή Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρη. Γενικώ η Αυστριακή Προεδρία διοργανώθηκε σωστά, ήταν αποτελεσματική και καλά συντονισμένη. Και αυτό γιατί η Αυστρία είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί εύρυθμα. Ε, καλύψατε πολλά θέματα στην ομιλία σας. Εγώ θα επιλέξω μόνο μερικά μεμονωμένα σημεία, ξεκινώντας με τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ήταν ε, σχεδόν διασκεδαστικό να ακούσουμε μια διαφορετική σκοπιά από την πλευρά της Προεδρίας και της Καγκελαρίας από ότι στο παρελθόν συνέβαινε. Είπατε ξεκάθαρα κάτι που άλλοι πολιτικοί δίσταζαν να πούν καθαρά, ότι η Ευρώπη δεν είναι ούτε έτοιμη ούτε πρόθυμη να δεχτεί ε, αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών. Ε, αυτό θα είχε επιπτώσεις και στην ασφαλεία μας, αλλά και στην εσωτερική μας συνοχή, στις κοινωνίες μας. Και επίσης ε, υποβάλλατε ε, προτάσεις και λύσεις, όπως την αναθεωρήση του κώδικα των συνόρων για το Σέγγεν και την ε, αρρωγή για την υποδοχή της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση της λάθρομετανάστευσης. Σίγουρα τα μηνύματά σας αυτά ακούστηκαν από πολλούς με προσοχή, ξεκάθαρα, και στην κεντρική Ευρώπη και σε άλλες χώρες και πάλι αποδείχθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναζητάτε συμβαστική λύση μεταξύ των κρατών μελών αντί να επιλέγουμε αυθαίρετες λύσεις, όπως ε, το ατυχές ε, σύστημα επανεγκατάστασης που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κόστισε μάλλον προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες διενέξεις μεταξύ Δύσης και Ανατολικής Ευρώπης και σίγουρα ε, έφερε ένα νέο διαχωρισμό μεταξύ κρατών και νέων και παλαιών κρατών μελών. Σίγουρα η ευημερία και η ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία είναι κάτι που προάγατε με την ψηφιοποίηση και την κοινοτομία και είχατε δίκιο ενώ λειτουργεί καλά η κουλτούρα μας για τις νοφείς επιχειρήσεις, ε, οι μεγάλοι στο χώρο αυτό έρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να άρουμε τους εμπορικούς φραγμούς και θέλω να σας συγχαρώ γιατί πετύχατε τη γρήγορη έγκριση της εμπορικής ε, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ιαπωνία. Έτσι δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη εμπορική περιοχή καλύπτοντας το, ε, ένα το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ελπίζουμε να προχωρήσουν οι συμφωνίες με την Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν επί τη Προεδρία σα θα συνεχιστούν. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή φτάνουν στο τέλος τη θητείας τους. Δεν θα πρέπει να αποφασίσουν εκ μέρου των 100 μελών ή ε, προδικάζοντα το τι θα κάνουν οι μελλοντικοί Επίτροποι. Για τι εξωτερικέ μα σχέσει. Δεν θα επεκταθώ Απλώς να δηλώσω ότι η Αυστρική Προεδρία είχε πραγματιστική προσέγγιση, δεν ε, ήταν θύμα ιδεολογιών και επεδίωξε χειροπιαστά και αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή η κοινή λογική ε, υπερίσχυσε. Ε, η κοινή λογική είναι και κάτι που προσπαθεί να προάγει και η δική μου η ομάδα σε αυτό το κοινοβούλιο. Επιτέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Τελίτσκα, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Καγκελάριε, δεν είμαι βέβαιος εάν θα αντέξετε να ακούσετε κι άλλα συγχαρητήρια, γιατί ακούσατε ήδη πολλά σήμερα, οπότε θα σας απαλλάξω. Ήταν αποτελεσματική η προεδρία σας. Η Αυστρία έφερε αποτελέσματα, ε, ήταν συνεπής με όσα είχε αρχικά ανακοινώσει, όμως κάθε έξι μήνες το θέμα δεν είναι αν τα πήγε καλά απλώ η Προεδρία. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε μόνο αυτό, αλλά και το πώ τα πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτω Προεδρία. Αυτό που πρέπει λοιπόν να ακουστεί σήμερα είναι ότι μιλάμε ακόμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, που μπορεί σύντομα να είναι 27 κράτη-μέλη. Η Προεδρία έχει το ρόλο τη να διαδραματίσει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη τη, αλλά μπορεί να κάνει πολλά για την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν ήδη είναι ένα ε, καλό Τώρα μιλήσατε για τον αριθμό των τριμερών διαλόγων και αυτό είναι ε, ένα δείγμα ε, αποτελεσματικής προεδρίας, αλλά να δούμε τι έγινε με την νομοθεσία που εφαρμόζεται. Είναι ε, η νομοθεσία που εγκρίθηκε αυτή που θα επιδιώξει τους στόχους που ανακοινώσατε και εσείς, τους τρεις στόχους που αναφέρατε προηγουμένως. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η συγγήτρια Αγγελικά ασχολήθηκε με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα, ήταν μάλλον καλό. Όμω, παρά τι διάφορε διαφιλονικίε που είχαμε με τον πρεσβευτή τη Αυστρία, ε, που είχε πολύ έντονη παρουσία στου τριμμένου διαλόγου, παρόλα αυτά αντικατοπτρίζεται η έλλειψη αλλαγή νοοτροπία και κουλτούρα στα κράτη-μέλη. Ακόμη την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τον την βλέπουν σαν ένα θέμα όπου παίζουμε ε, μεταξύ όσων θέλουν ε, να προασπιστούν εταιρικά συμφέροντα και όσων όχι. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε δυνατοί ή αδύναμοι. Είμαστε ο πιο δύναμο κρίκο τη αλυσίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω το εξή. Ε, το, θέμα δεν είναι απλώ πόσου τριμμένου διαλόγου ε, οργανώσαμε, αλλά τι νομοθεσία εγκρίναμε και τι κατάφεραν να συμφωνήσουν μεταξύ του τα κάθε μέλη με συμβαστικέ λύσει για το επίπεδο φιλοδοξιών του. Για την ε, ψηφιακή προστασία των δεδομένων. Ε, ναι, υπήρξε πρόοδος, αλλά εγώ αν είχα το μυαλό θα μπορούσα να εφεύρω μια ε, εφαρμογή που να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να την πουλήσω εγώ στο Silicon Valley. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Δυστυχώ δεν έχω το μυαλό. Είναι πολλά λοιπόν που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπορικό τη οικοσύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε δύο-τρία ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Οπωσδήποτε και είναι και ένας γνώμονας για την Προεδρία. Το ένα είναι η ε, εσωτερική ασφάλεια. Ναι, είχατε καλά εξισορροπημένη προσέγγιση, όμως δεν το παραδεχτούμε. Ακόμη έχουμε μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο για πολλέ προτάσει οι οποίε εκκρεμούν. Είναι σε τέλμα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κρίση και τα τωρινά προβλήματα ε, με αυτέ τι λύσει. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα αν αυτά ενταθούν για τον προπολογισμό. Και πάλι Τεράστια πρόοδο επετέχθη, δεν μπορώ να πω. Όλα τα κουτάκια που έπρεπε να συμπληρώσετε πήραν τικ. Αλλά πώ συμπληρώθηκαν. Όπω είπε ο κύριο ε, Ζάχραντιλ, ε, να τα αφήσουμε αυτό στην επόμενη θητεία. Όχι, ε, εξελέγημεν, για ολόκληρη τη θητεία εμεί, για την ολόκληρη την πενταετία. Άρα, όταν μιλάμε για την συνοχή, αν μιλάμε για του γεωργού και βλέπουμε ότι καθυστερούμε, αυτό επηρεάζει τι δουλειέ του, επηρεάζει το πώ θα πάνε. Οπότε ο προπολογισμό είναι ένα δείγμα για το πώ ε, μα αντιλαμβάνονται απ' έξω. Και δεν είναι κατηγορία για την Αυστρία αυτό. Είσαστε ρεαλιστέ, ναι, και εγώ είμαι κατά τη οποιασδήποτε σπατάλη και διασπάθηση ε, κονδυλίων. Όμω με τι νέε προκλήσει που έχουμε μπροστά μα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε απλώ να αναθεωρούμε κάποιε πολιτικέ και ε, να μην αυξάνουμε πουθενά τον προπολογισμό. Και εν τέλει, με αυτέ τι παρατηρήσει, παρόλα αυτά να πω ότι η δουλειά σα ήταν καλή, αλλά ω Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν είμαστε στο ύψο των προσδοκιών των συμπολιτών μα σε πολλά ζητήματα μένουμε πίσω. Ευχαριστώ. Τώρα, στην κυρία Σκακέλερ από τους Πρασίνους θα δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δυστυχώ. κύριε Κούρτς δεν μπορώ να συνταχθώ με τους ε, προλαλήσαντες. Τι απέμεινε τελικά από την Αυστριακή Προεδρία δεν προχώρησαν. Πολλές νομοθετικές προτάσεις κόλλησαν στο Συμβούλιο, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά θα μας μείνει σε εμά και εκτός από την αίθουσα στους τελευταίους έξι μήνες είναι η πραγματικά λυπηρή υπόκλησή σας στον πρόεδρο Πούτιν. Αλλά και το ότι αρνηθήκατε να συνυπογράψετε το σύμφωνο του ΟΗΕ για την μετανάστευση ειδικά η αυστριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει αυτή την προσπάθεια τόσων πολλών κρατών του κόσμου για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά ενώ καταβάλατε κι εσείς προσπάθεια στο να συνταχθεί, να παριστάνετε μετά ότι είναι του σατανά, είναι ανεξήγητο. Ε, Πολώσατε λοιπόν και μπήκατε μόνοι σας ε, στην ε, ακροδεξιά γωνία όπως ο Τραμπ και ο Όρμπαν. Και εκεί πέρα μας βλάψατε όλους, ε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι έτσι. Ξεκαθαρό ότι η κυβέρνησή σας έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε ενώ υπήρχε διακριτική μεταχείριση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το να περικοπούν κάποια οικογενειακά βοηθήματα. Τέλος πάντων. Στα θετικά όμως ε, δεν υπάρχουν τόσα πολλά στους τελευταίους ε, έξι μήνες ούτε στην καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής και του φορολογικού dumping ούτε σε ζητήματα διοξιδίου του άνθρακα. Εκεί πέρα απλά ήσασταν ε, παρακολούθημα της ε, γερμανικής ε, αυτοκίνητοβιομηχανίας. Δεν έγινε και τίποτα και στην Frontex. Ούτε καν στην Frontex αναβλήθηκαν τα πάντα και υποτίθεται ότι ήταν προτεραιότητα της Αυστριακής Προεδρίας. Όσον αφορά όντως τα πλαστικά μιας χρήσης κάτι έγινε και εδώ πέρα πρέπει να επενέσω τους υπαλλήλους σας και νομίζω ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση της ε, Προεδρίας σας ε, ήταν ε, ότι κερδίσατε στο Κατοβίτσε το βραβείο που δώσαμε για το απολύθωμα της ημέρας. Αλλά η κοινωνία των πολιτών στην Αυστρία είναι διαφορετική. Πάρα πολλοί κόσμος εμπλέκεται, βγαίνει στους δρόμους κατά του ρατσισμού και κατά της μείωσης του κοινωνικού κράτους και ελπίζω ε, να κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι στην Αυστρία και στις ε, ευρωεκλογές γιατί η Ευρώπη χρειάζεται μια Αυστρία ανοιχτή στον κόσμο και ολόκληρη η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινωνία των πολιτών όπως η δική σας ε, κατά του διχασμού και υπέρ της κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ, ο κύριος Παπαδημούλης έχει το λόγο. Κύριε Κούρτς, λυπάμαι, αλλά θα σας απογοητεύσω. Δεν συμμερίζομαι το κλίμα των αυτοεπένων και των συγχαρητηρίων. Θεωρώ ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Αυστρία ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκε να υπογράψει το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση στο Μαρακές. Ένα σύμφωνο που υπέγραψαν 150 χώρες από όλο τον πλανήτη μετριοπαθές, ισορροπημένο, στην προετοιμασία του οποίου είχατε συμβάλει. Και θέλω να μας απαντήσετε στη δευτερολογία σας. Γιατί ντροπιάσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προεδρεύων αρνούμενος να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτό το κείμενο. Δεν σας τα λέω μόνο εγώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Σας τα είπε πιο ευγενικά, πιο κομψά και ο κύριος Γιούνκερ που ανήκει στην πολιτική σας ομάδα. Και επίσης, δεν κάνατε τίποτα για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Δεν κάνατε τίποτα ουσιαστικό για να προωθήσετε το πακέτο μεταρρύθμισης του Δουβλίνου, στο οποίο έχουμε συμφωνήσει εδώ και καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Το καθυστερείτε και το μπλοκάρετε. Για την πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, το περίφημο EDIS, και πάλι αναβλητικότητα και καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η τραπεζική ενοποίηση. Για την φορολόγηση των γιγάντων του διαδικτύου. Τίποτα συγκεκριμένο. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δουλειά σας ήταν να επιταχύνετε τις συγκλήσεις για να έχουμε μια συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί η αναβολή λήψης αποφάσεων σε αυτό το θέμα κάνει ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πολύ φοβούμε ότι η συγκυβέρνησή σας με ένα κόμμα της άκρας δεξιάς, το οποίο ιδρύθηκε από οπαδούς των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σας επηρεάζει καθοριστικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τις ευρωεκλογέ μια τέτοια συμμαχία δεξιά άκρα δεξιάς. Επειδή σα επέκρινα πολύ, θα κλείσω με μια θετική αναφορά. Θεωρώ θετικό ότι και εσείς και ομόφωνα το Συμβούλιο και ομόφωνα η Κομισιόν και όλες οι πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια συμφωνία θετική για την Ελλάδα, θετική για τη Βόρεια Μακεδονία, θετική για τα Βαλκάνια, θετική για όλη την Ευρώπη είναι μία από τις καλές ειδήσει που έχουμε δυστυχώς λίγες αυτή την περίοδο και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τις επόμενες ημέρες η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι αποφασισμένη να κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών στο Κοινοβούλιο της Αθήνας παρά την αντίδραση, την μικροπολιτική την δημαγωγική των κομμάτων της νέας δημοκρατίας και του πασόκ που σε αντίθεση με τις πολιτικές ομάδες του ελκ και των σοσιαλιστών αντιπολιτεύονται και αρνούνται την κύρωση της συμφωνίας των πρεσπών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Άμεσης Δημοκρατίας ο κύριος Μόιτεν. Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Κούλτς. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω τρία θετικά πράγματα στα πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, η γη συνεχίζει να γυρίζει. Δεύτερον, δεν έγιναν πόλεμοι. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να γραφειοκρατικοποιείται. Και όλα αυτά παρά την πρεμιέρα αυτή που είχαμε. Οι λεγόμενοι δεξιοί λαϊκιστές συμμετείχαν για πρώτη φορά σε μια κυβέρνηση και αυτή είχε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό δείχνει πω κάποια πράγματα αλλάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα δραστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι ήταν πριν από την Αυστριακή Προεδρία. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο συνέβη για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά η Προεδρία του Συμβουλίου δεν ε, αισθάνθηκε την ανάγκη να είναι η πιο συγκεντρωτική ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ρεαλιστική, Χωρί να προωθεί τον συγκεντρωτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Εμεί το ΕΦΤΕ θέσαμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και τολμώ να ισχυριστώ ότι δεν θα είχε κυριαρχήσει στη συζήτηση στην Ευρώπη εάν δεν υπήρχε η αυστριακή κυβέρνηση η οποία ήταν πραγματικά αποφασισμένη και στις δηλώσεις της. Η Αυστρία πραγματικά κατάφερε να ξεχωρίσει από τους yes και έτσι κατάφερε να υπάρξει μια δημόσια συζήτηση για αυτό το καταστροφικό σύμφωνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Κούρτ. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Αυστριακή Προεδρία μία μέρα θα θεωρηθεί ένα σημείο καμπής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής ενωση Δεν είμαι ο μόνος, νομίζω, ο οποίος αντιλαμβάνεται την δύναμη που έχει μία Προεδρία του Συμβουλίου. είμαι σίγουρος ότι Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες προεδρίες του Συμβουλίου, το αυστριακό παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι, μια μικρή αντίσταση κατά της ε, ακόμα κυρίαρχης τάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σας καθιστά αντιευρωπαίους. Αντιθέτως, το να μην είστε γεσμεν και να λέτε συνεχώς αμήν και οσανά είναι υποχρέωση των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε επιτέλους κάποιες δικλείδες ασφαλείας που θα λειτουργούν, να ακουστεί και κάποιο όχι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπό την ηγεσία Κομισιών και Κοινοβουλίου λειτουργεί ως υπερκράτος. Αυτό το όχι θα το ακούμε συχνότερα στο μέλλον και θα κάνει καλό στην Ευρώπη. Αυτό προβλέπω εγώ. Ευχαριστώ. Την Ευρώπη των Εθνών και ε, των Ελευθεριών, ο ε, συνάδελφε Ελίνσκι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σαν Αυστριακός θα ήθελα να ξεκινήσω ευχόμενος στον καγκελάριό μας, τον κύριο Σεμπάστιαν Κόλτς, καθώς ήρθε, το καλώς ήρθε στο Κοινοβούλιο και στον κύριο Κούρτς και θα ήθελα να διαβιβάσει ευχαριστήσεις στην αντιπροσωπεία μου ε, και να διαβιβαστούν αυτέ οι ευχαριστήσει και προ την κυβέρνηση. Αυτή η Προεδρία του Συμβουλίου, η Αυστριακή, ήταν πολύ επαγγελματική, πάρα πολύ επαγγελματική και υποδειγματική για όλους εκείνους που προσπαθούν να κατηγορήσουν ή να αναμαυρώσουν την Αυστριακή Προεδρία, πρέπει να πω ότι πρέπει να πούμε στους σοσιαλδημοκράτες ότι έχουμε και, έχετε τους Ρουμάνους σοσιαλδημοκράτες στην ομάδα σας και πρέπει να το θυμηθείτε αυτό. Και αν βλέπετε τα θέματα διαφθοράς και άλλα συναφή θέματα, να θυμηθείτε ότι δεν είσαστε ε, ε, και πολύ δεν είσαστε τόσο αθώοι ώστε να κατηγορείτε άλλους. Και οι πράσινοι συνεχώς διαμαρτύρονται για το κόμμα ελευθεριών, ε, της ελευθερίας στην Αυστρία. Αλλά εκείνο αποφάσισε, αυτό το κόμμα αποφάσισε στην Αυστρία να εργαστεί σκληρά για το θέμα των αποζημιώσεων και τη συνεργασία με το Ισραήλ. πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να μην ε, απαγγέλουμε κατηγορίες κατά άλλων κομμάτων. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί η Αυστρία δεν επικύρωσε ε, το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Διότι υπήρχε μια τέτοια δημοκρατική πλειοψηφία εντός της κυβερνήσεως και του Κοινοβουλίου που ήθελε να συνεχίσουμε να καθορίζουμε εμείς τη μεταναστευτική μας πολιτική, εμείς οι ίδιοι και δεν θέλαμε να κυρώσουμε ένα μη δεσμευτικό σύμφωνο που τελικά θα κατέληγε από μη δεσμευτικό να καταλήξει, θα γινόταν δεσμευτικό. Νομίζω ότι είναι σωστό να μην αγνοήσουμε και τη θέση του ανωτά του δικαστηρίου μας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Αυστρίας στο Συμβουλίο, το θέμα της επικουρικότητας ε, στηρίχθηκε δεόντω. Έγινε μια διάσκεψη στο Μπρέγκενς όπου άνοιξε το δρόμο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έλεγε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε εθνικές αποφάσεις και είναι καλύτερο να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η Προεδρία του Συμβουλίου η Αυστριακή υπήρξε έξοχη και ελπίζω ότι μια τέτοιου είδους Προεδρία θα είναι υπόδειγμα για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αστική κυβέρνηση. Το έχει ο κύριο Ουγιασδόφσκι από του Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καγκελάριο κύριο κουρτ για την πολύ ρεαλιστική και πραγματιστική Αυστριακή Προεδρία που άσκησε. Γιατί είναι πολύ πιο θετική αυτή η στρατηγική γευνακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στρατηγική της περισσότερης ολοκλήρωσης και της πιο περισσότερης και πιο παρούσης Ευρώπης. Ιδιαίτερα στα θέματα της οικολογίας, της προστασίας, της αγοράς απέναντι στα μεγαθύρια του ίντερνετ. Ήταν πολύ σημαντικά επιτεύγματα της Αυστριακής Προεδρίας. Τα παρουσιάσατε και στην ομιλία σας. Μάλιστα υπήρξε μεγάλη διαφορά με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική. Και αυτέ οι διαφορέ μεταξύ ε, Κομισιόν και Συμβουλίου δείχνει πόσο πιο λογική ήταν η Αυστριακή Προεδρία, γιατί η αλληλέγγυα πολιτική απέναντι στου μετανάστες θα πρέπει να είναι υπεύθυνη πολιτική και ρεαλιστική πολιτική, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διέπραξε μείζον σφάλμα ε, επιβάλλοντας το σύστημα των ποσοστώσεων για την υποδοχή μεταναστών κάτι που μείωσε την εμπιστοσύνη του λαού προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οδήγησε σε μια αύξηση και σε έξαρση του λαϊκισμού, της δημαγωγίας. Ε, θα πρέπει να είμαστε συνετοί, σόφρονες, να ασκούμε μια αλληλέγγυα πολιτική που θα είναι όμως πρώτα απ' όλα ρεαλιστική. Και καλό θα ήταν να αναλογιστούμε την πολύ θετική εμπειρία της Αυστριακής Προεδρίας από την άποψη αυτή. Επίσης, ε, συμφωνώ να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, όπως είπε ο καγκελάριος Κούρτς, και πιστεύω ότι θα ε, τεθούν σωστά θεμέλια, ώστε να γίνει μια ευαισθητοποίηση υπέρ της ανεξιθρησκείας και της ελευθερίας της ε, θρησκευτικής πεποίθησης. Και κυρίως να προστατεύσουμε τους χριστιανούς, που είναι η θρησκευτική ομάδα στον κόσμο που κατεξοχήν διώκεται. Ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ζων Κλοντ Γιούγκερ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι ε, που έχω να προσθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω απλώς την Αυστριακή Προεδρία και σε ό,τι αφορά αυτά που υπόθηκαν για την μετανάστευση και την πολιτική της Αυστριακής Προεδρίας. Εγώ μιλώ όχι μόνο εξ ονόματός μου, αλλά και εξ ονόματος ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής συνολικά. Και όσοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν ανήκουν σε μια δημοκρατική συζήτηση, πλανώνται. Πάντως έχω να πω ότι υπήρξε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα της Αυστριακής Προεδρίας. Και μπορούμε να πούμε ότι στην ε, σύντομη ιστορία των Προεδριών της Ένωσης η Αυστριακή Προεδρία θα μείνει σαν μία από τις πιο επιτυχημένες και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Τώρα ε, ε, Αξιότιμε κύριε πρόεδρε Ταγιάννη, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Δεν μου μένουν πολλά να πω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θετικά λόγια σας σήμερα. πραγματικά υπάρχει συμφωνία που μας ενώνει σε πολλούς σημαντικούς τομείς ε, και πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τις ακούσαμε, αλλά και μεταξύ των ομάδων να εκπροσωπούνται διαφορετικές απόψεις. Ε, Αυτό είναι το οποίο διαμορφώνει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Παρά όμως τις διαφορές και τις ενδεχόμενες διαφωνίες, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε από κοινού και να προβούμε στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσει, τι οποίε θεωρούμε ότι είναι σημαντικές. Ε, 28 κράτη-μέλη, τρία θεσμικά όργανα πολύπλοκα και η συνεργασία πολύπλοκη. Είμαι σίγουρη ότι καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε 53 τριμερείς διαλόγους και νομίζω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Συμβούλου καταφέραμε να καταλήξουμε σε ομοφωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ρουμανική Προεδρία που παίρνει τη σκητάλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δέσμευση αυτή που αναλάβατε και την προσπάθεια. Διακόπτουμε για μερικά λεπτά τη συνεδρίαση. Πριν την πανηγυρική συνεδρίαση για την 20η επέτειο του ευρώ.